μια μεγάλη πρόοδο για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο για τα καλά του λόγια, ευχαριστώ τους συναδέλφους και τους ε, συναδέλφους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συζήτηση περατώθηκε, η ψηφοφορία θα δεξαχθεί αύριο στις 12.30 το μεσημέρι. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή και αφορά την νομική κατάρτιση εξ ονόματος της Επιτροπής νομικών θεμάτων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Συντάκτης, ε, δίνω το λόγο στον, σε έναν εκ των συντακτών, στον κύριο Ζεύκα Ταντέους, για δύο, δύο, για δύο μισή λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Στη Νομική Επιτροπή Φυσικό είναι καθημερινά να ε, ε, εξετάζουμε διάφορα νομοθετικά κείμενα σε ό,τι αφορά το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο διαδοχής, το εμπορικό δίκαιο και πρέπει να πω ότι όταν αυτά τα σχέδια θα, θα καταστούν υποχρεωτικοί νόμοι θα απαιτήσουν από τους δικαστές ιδιαίτερες γνώσεις όχι μόνο για το δικό τους δίκαιο, αλλά και το δίκαιο που ισχύει στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς δουλεύουμε στα πλαίσια της νομικής μας επιτροπής, σε συνεργασία με τον Λουίτζι Μπέρλιγκερ συζητήσαμε πολύ για το θέμα της κατάρτισης που πρέπει να έχουν οι τα διάφορα άτομα που θα κληθούν να εφαρμόσουν αυτές τις διατάξεις. Θα υπάρχουν όλο και πιο συχνά ε, ανάγκες για τέτοιες γνώσεις εξειδικευμένες διότι αυτά θα είναι θέματα που θα μας αφορούν όλο, όλους. Οι διατάξεις αλλάζουν καθημερινά. Χρειάζεται λοιπόν ε, ιδιαίτερη επιμέλεια από πλευράς των δικαστών και των άλλων νομικών η κατάρτιση αυτών των λειτουργών αφορά το ολόκληρο το σύστημα της δικαιοσύνης και πρέπει να έχουμε πείγνωση των προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουμε και που θα χρειαστεί να λύσουμε. Αυτή λοιπόν η κατάρτιση είναι απολύτως αναγκαία, απολύτως απαραίτητη. στους συναδέρφους λένε και Λόπες Αγγιλάρ θέλουμε να εκφράσουμε την ανησυχία μας για αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα που έχει σκοπό να προσφέρει την αναγκαία κατάρτιση στο ίμιση τουλάχιστον των δικαστών και των άλλων λειτουργών και υπαλλήλων του τομέα απονομής της δικαιοσύνης ώστε ε, ποιο θα είναι το πλαίσιο ανταλλαγή εμπειριών, σε τι ποσοστό θα μπορέσει να συμμετάσχει σε αυτή τη σημαντική εργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Από την αρχή της εφαρμογής του προγράμματος της Στοκχόλμης μιλάμε για την ανάγκη μιας ευρωπαϊκής νομικής κουλτούρας. Όλα τα θεσμικά όργανα τα ευρωπαϊκά, ενώ υποστηρίζουν αυτό το πρόγραμμα, αντιλαμβάνονται ότι αυτή η ακατάρτιση είναι αναγκαία. Σχετικά με το πρόγραμμα Δικαιοσύνη για το 2014-2020, το θέμα της κατάρτισης είναι ιδιαίτερα σημαντικό ώστε να μπορέσουμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά μεταξύ μας. Χρειαζόμαστε, χρειάζεται να μπορούμε να χρησιμοποιούμε μια κοινή γλώσσα. Χρειάζονται λοιπόν ε, προγράμματα επιμόρφωσης και ειδικά προγράμματα στις νομικές σχολές των, ε, των ε, Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Όπως είπε ο συνάδελφος Γεύκα, θα θέλαμε το θέμα αυτό να οδηγήσει σε συζήτηση. Μιλάμε λοιπόν για την ε, νομική κατάρτιση, για την κατάρτιση νομικών που εφαρμόζουν καταρχήν το κοινοτικό δίκαιο. Μιλάμε για ε, ένα νομικό οικοδόμημα και γι' αυτό ακριβώς έχουμε επιτύχει αυτό το είδαμε από τις συνθήκες του Άμστερνταμ, της Νίκιας και στη συνέχεια της Λισαβόνας. Μιλάμε λοιπόν για, μεγάλες, για μια μεγάλη ανελικτική πορεία τα τελευταία δέκα χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν οι δικαστικές αρχές, οι δικαστές και οι εισαγγελείς να έχουν την κατάλληλη κατάρτιση με βάση την ένομη τάξη των κρατών μελών έτσι ώστε να μπορούν να αποφανθούν. Θα πρέπει παράλληλα να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο φορέων νομικής κατάρτισης έτσι ώστε να υπάρχει μία συνέργεια με την Κομισιόν και γι' αυτό θα θέλαμε να ξέρουμε πώς προβλέπει η Επιτροπή να επιτύχει με βάση προσφορές κατάρτισης μέχρι το 2020. Δεύτερον, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με το δίκτυο φορέων νομικής κατάρτισης. Τρίτον, πώς θα ενισχύσει η Επιτροπή το ρόλο των φορέων και δικτύων για να δώσει μία νέα όθηση σε αυτό το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και πώς θα ε, οργανωθεί το προτινόμενο πιλωτικό έργο για την κατάρτιση δικαστών και εισαγγελέων. Μιλάμε για τον μεγάλο καταλήτη συνεργασίας μαζί με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζονται το ίδιο όραμα για αυτό το θέμα και χάρη στη συνεργασία ανάμεσα στην Επιτροπή, την Νομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ελευθεριών έχουμε ένα ψήφισμα που αναφορά την ανακοίνωση που ενέκρινε η Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Νομική Κατάρτιση το Σεπτέμβριο του 2011. Αυτό που θα ήθελε να κάνει η Επιτροπή είναι να δώσει όθηση σε ένα νέο χώρο δικαιοσύνης, δημιουργώντας ένα νέο χώρο δικαιοσύνης που θα εμπνέει εμπιστοσύνη και για να γίνει αυτό η κατάσταση των νομικών πρέπει να ενισχυθεί. Έχουμε θέσει ως στόχο 700.000 ε, λειτουργοί δικαστικών λειτουργών στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν συμμετάσχει σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης ε, για το Ευρωπαϊκό Δίκαιο μέχρι το 2020. Για να επιτευχθεί αυτός ο φιλόδοξος αλλά και ρεαλιστικός παράλληλα στόχος, όλοι οι διαθέσιμοι πόροι σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο θα χρειαστεί να αξιοποιηθούν και να κινητοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν και βεβαίως όλες οι ενδιαφερ... τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να δεσμευθούν να εντάξουν το ενωσιακό δίκαιο και, ε, την εφαρμογή του μέσα από προγράμματα κατάρτισης, να αυξήσουν αυτά τα προγράμματα κατάρτισης για το ευρωπαϊκό δίκαιο και τον ρυθμό ε, ε, των ατόμων που θα συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα. Επίσης, με, με βέλτιστο τρόπο πρέπει να οργανωθεί αυτή η κατάρτιση ώστε ε, να, ε, τα προγράμματα αυτά να είναι πραγματικά αποτελεσματικά. Βεβαίως θα συνεργαστεί με, τις, με, με τα ενδιαφερόμενα μέρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου, το, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημοσίου Δικαίου. Θα συνεργαστεί επίσης στενά με τους ε, επαγγελματικές νομικές οργανώσεις. Επίσης θέλουμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα ανταλλαγών δύο εβδομάδων για ε, εισαγγελείς και δικαστές από το 2014 και πέρα και δεσμευόμαστε να θέσουμε ε, τα απαραίτητα κονδύλια, να είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα κονδύλια για την χρηματοδότηση σημαντικών προγραμμάτων σε ό,τι αφορά τη συνέχεια στο πιλωτικό πρόγραμμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα ώστε να υπάρξει αρχές της Άνοιξης μια ευρωπαϊκή απόφαση. Ο κύριος Γιακολίνο τώρα για δύο λεπτά από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και την Επίτροπο. Ακούσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις υποδείξεις της Επιτροπής για την προώθηση της νομικής κατάρτισης. Θεωρούμε ότι είναι θέμα ύψης της ε, σημασίας γιατί θα πρέπει να δούμε πώς έχουν οι διάφορες ένομες τάξεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η συγκεκριμένη συνεργασία η οποία θα μπορούσε να διευκολύνει την διακρατική συνεργασία. Θα πρέπει ο δικαστικός μηχανισμός να είναι ενιαίος, να την χάνει ενιαίας πρικοδότησης και κατάρτισης και μέσω του Εράσμους, έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη και την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα. Όλα αυτά συνδέονται με την απελευθέρωση των επαγγελμάτων, κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία για τις διάφορες προδιαγραφές και εχέγγυα επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτό μας ορίζει και το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Μιλάμε για την αμοιβαία αναγνώριση των διαφόρων νομικών πλαισίων και αυτό αφορά μια ενιαία αγορά εργασίας γιατί μας ενδιαφέρει να μπορούμε να χρησιμοποιούμε και όσο το δυνατόν περισσότερες γλώσσες. Οι δημοσιονομικές προοπτικές 14-20 θα πρέπει να ε, διέπονται από συγκεκριμένες αρχές και να υπάρχουν και οι κατάλληλοι πόροι έτσι ώστε να υπάρχει μια ευρεία πλατφόρμα νομικής κατάρτισης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα εν ονόματι των σοσιαλιστών ο κύριος Μπερλίνγκουερ. Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε σε σωρία νόμων, κανόνων και ούτω καθεξής για την οικοδόμηση του κοινοτικού δικαίου και έφτασε στον ευρωπαϊκό χώρο επωνόματι πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Μιλάμε για ένα νομοθετικό κόρπους που έχει μεγάλη σημασία για τους πολίτες. Απ' την άλλη πλευρά, οι εθνικοί δικαστές ασχολήθηκαν με το ε, δίκαιο της χώρας τους ενώ εμείς θεωρούμε ότι ο πραγματικός Ευρωπαίος δικαστής είναι ο εθνικός δικαστής ο οποίος αλλάζει ρόλους. Δηλαδή διέπεται από ε, μία διάθεση επικοινωνίας προς τους πολίτες για να μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τα πλεονεκτήματα αυτού του δικαίου. Πρόκειται για μία κίνηση από τα κάτω προς τα πάνω. Δεν κάνουμε μαθήματα όπως κάνουμε στην ε, πρώτη δημοτικού. Θα πρέπει να μπορούμε να συσχετιζόμαστε με τους ε, άλλους συναδέλφους, διότι common law και civil law συγκλίνουν, δεν ε, αποκλίνουν όπως ίσχυε κάποτε. Χαίρομαι διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίστηκε για αυτό, το, για αυτή την προσέγγιση bottom-up δηλαδή, από τα κάτω προς τα πάνω. Υπάρχει το Eurinfra στην Ολλανδία. Είναι ένα δίκτυο πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή κάθε δικαστήριο δίνει τα φώτα του στις δικαστικές αρχές. Ελπίζουμε να μας υποστηρίξει η Επιτροπή σε αυτό μας το εγχείρημα. Ευχαριστώ. Εν ονόματι των φιλελευθέρων, η Σεσίλια Βίξτρα με έχει το λόγο τώρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην ε, ε, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα υπάρχει κατανόηση ότι όλοι διαφέρουμε μεταξύ μας και πλέον Είμαστε ενωμένοι στην πολυμορφία μας, πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την ολοκλήρωση της Ευρώπης. Πρέπει να σκεφτούμε από κοινού πώς θα μπορέσουμε να βρούμε ε, κοινά τρόπους για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την κοινή πορεία μας, γιατί μόνο με ανταλλαγή απόψεων θα μπορέσουμε ε, να προσεγγίσουμε παρά τις διαφορές μας και να υπάρξει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Είμαι πεπισμένη ότι αυτό ισχύει και για τα νομικά επαγγέλματα, για τους δικαστές, ε, για τους συμβολογράφους, για τους νομικούς και είναι βασικό να μπορούν να συνεννοούνται όταν θα συναντιούνται και θα μπορούν να ανταλλάσσουν απόψη, να καταρτήσουν κάποιο διάλογο και να μπορέσουν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον να να εξελιχθούν και περαιτέρω μέσω αυτής της συνομιλίας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει μία συνεννόηση και θα επιλύσουμε τα θέματα των διαφορών. Βεβαίως θα πρέπει να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη και όλες τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ κρατών μελών και να φροντίσουμε να υπάρξει μία αμοιβαία νομοθεσία η οποία θα πρέπει να γίνει κατανοητή ε, κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να προοδεύσουμε και να μπορέσουμε να συμβάλλουμε εις ε, την ε, πρόθεση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ευχαριστώ που σεβαστήκατε το χρόνο σας και τώρα θα δώσω για ένα λεπτό τον λόγο στον κύριο Ανδρέας Μέλτσερ. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μία πληθώρα όχι μόνο εθνικών νομοθετημάτων αλλά και ευρωπαϊκών νομοθετημάτων που επηρεάζονται από το διεθνές δίκαιο και επιπλέον συνεχείς νομικές εξελίξεις. Για να μπορεί κανείς να αντεπεξέλθει σε αυτές τις εξελίξεις χρειάζεται η επιμόρφωση η οποία είναι απαραίτητη και μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει κανείς να ενισχύσει την προστασία των θυμάτων διότι ε, γι' αυτό το λόγο και μόνο ε, είναι απαραίτητη η περαιτέρω εξέλιξη του ε, νομικής επιστήμης και των δικαστών κατά τρόπον ώστε να μπορέσουν να υπερασπιστούν τα θύματα διακρίσεων και ε, ε, θα πρέπει βάσει της ε, διακηρύξεως υπαριθμών 34 του ΟΗΕ να δούμε ότι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη υπάρχουν πολλές νομοθεσίες οι οποίες ποινικοποιούν παραδείγματος χάρη τη γενοκτονία των Αρμενίων οι οποίες θα πρέπει να επιληθούν σε διεθνές επίπεδο. Σας ευχαριστώ. Πλέον ερχόμαστε στις, ε, στους άλλους ομιλητές, στην Ερμίνα Ματσόνη από το ΕΛΚ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο Ρέντινγκ για την σημαντική της εργασία σε αυτό το ε, πολύ σημαντικό ζήτημα, δηλαδή να δώσει σάρκα και οστά σε αυτό το εγχείρημα νομικής ε, κατάρτισης. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπέρλιγκουέρ, ο οποίος ε, μας δίνει τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα της Στοκχόλμης μετά την τελευταία ανακοίνωση της Επιτροπής του Σεπτεμβρίου, στην οποία αναφέρθηκε η Επίτροπος Ρέντινγκ ο στόχος του πιλωτικού σχεδίου, όπως είπε ο κύριος Μπερλιγκουέρ, ορίζει μια κοινή πλατφόρμα δικαίου όπου υπερβαίνουμε τις δυσκολίες και μεταξύ επαγγελμάτων και όχι μόνο κρατών υπάρχουν καινοτόμα στοιχεία τα οποία κρίναμε ότι θα πρέπει να εισαγάγουμε σε αυτό το σχέδιο. Δεν μιλάμε για την συνεχή κατάρτιση, όπως είπε ο κύριος Μπερλιγκουέρ, αλλά θα πρέπει οι συμβολεογράφοι, οι δικαστές, οι δικηγόροι, οι να συμμετέχουν σε αυτό το κοινό εγχείρημα κατάρτισης. Η κυρία Ρέντινγκ είπε πολύ σωστά ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο εκκίνησης. Όμως η κυρία Ρέντινγκ δεν μας έκανε αρκετές υποδείξεις σε σχέση με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για αυτό το πιλωτικό σχέδιο. Θα πρέπει ένα πειραματικό σχέδιο να σε αυτό το σχέδιο να συμμετέχουν όλοι οι φορείς και όχι μόνο οι δικαστικοί. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή να μπορέσουμε να συμμεριστούμε μία κοινή βάση αποκλειστικά εμείς, αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έτσι ώστε το πρωτόκολλο της Στοκχόλμης να φτάσει στον απότερο στόχο του. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκιόντς έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, της, ε, στην κοινή αγορά είναι βασικό να υπάρχει κινητικότητα και των κεφαλαίων και των ατόμων υπάρχουν όλο και στενότερες σχέσεις και προσωπικές και επαγγελματικές πράγμα το οποίο σημαίνει ότι και οι διαφορές θα πρέπει να επιλύονται υπάρχουν όλο και περισσότερο διασυνοριακές διαφορές πράγμα το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει κοινή αντιμετώπιση του ευρωπαϊκού δικαίου είναι προϋπόθεση της κινητικότητας οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη ε, ε, στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια διότι ε, θα πρέπει οι δικαστές να γνωρίζουν καλύτερα το ευρωπαϊκό δίκαιο και σαν σκιώδης εισηγήτρια του προγράμματος Justice από το 2014 στο 2020 θεωρώ απαραίτητο να μπορέσουμε να επιμορφώσουμε τους Ευρωπαίους δικαστές και εισαγγελείς διότι δεν θα πρέπει, να, θα πρέπει όλοι να μπορούν να ελέγχουν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η κυρία Ρέγνερ είναι η επόμενη ομιλήτρια για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία η Η ε, η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει αποδώσει ένα κονδύλι για την περαιτέρω επιμόρφωση των δικαστικών και νομικών κατά τρόπον ώστε ε, να μπορέσουν να αξιοποιηθούν οι εθνικές και κοινοτικές δυνατότητες επιμορφώσεως. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι πώς θα επιλύσετε τον γλωσσικό φραγμό, το γεγονός γεγονός ότι πολλοί δικαστές δεν γνωρίζουν ξένες γλώσσες και θα πρέπει να παρακολουθήσουν ε, διεθνή προγράμματα. Πώς λοιπόν πρόκειται ε, εσείς να εφαρμόσετε ε, την, το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο δίνει καλές ιδέες για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν βίντεο συνεδρία κατά τρόπον ώστε να μπορέσουν ε, και με άλλα μέτρα να εξοικονομηθούν κεφάλαια διότι επιπλέον οι δικαστικοί και οι δικαστές πρέπει να εμπλακούν οι ίδιοι γιατί γνωρίζουν καλύτερα ποια είναι τα προβλήματά τους και πώς θα μπορέσουν να επιληθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα ερχόμαστε στη δικασία Catch the ο κύριος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να καταθέσω μια, μια πραγματική προσωπική εμπειρία. Διατελώντα κάποια στιγμή συνήγορο υπεράσπιση στη χώρα μου στην Ελλάδα ενός φυσικού προσώπου, επικαλέστηκα το Ευρωπαϊκό Δίκαιο συγκεκριμένες διατάξεις προκειμένου να στοιχειοθετήσω την υπεράσπιση του συμπολίτη μου ο δικαστή τότε αναγκάστηκε να διακόψει και μάλιστα να αναβάλει την υπόθεση για κάποιους μήνες ώσπου δηλαδή να λάβει ερμηνεία από το ευρωπαϊκό δικαστήριο για ένα ζήτημα το οποίο ήταν συγκεκριμένο δυστυχώς όμως δεν υπήρχε η εμπειρία η εξοικείωση του εθνικού δικαστή να κριθεί απευθείας ως επίδικο ζήτημα τη στιγμή της δίκης. Και νομίζω αυτά τα παραδείγματα τα συναντούμε συχνά σε πολλά κράτη-μέλη. Το αποτέλεσμά τους είναι περισσότερη ταλαιπωρία για τους πολίτες, μεγαλύτερη γραφειοκρατία και καθυστέρηση στον χρόνο εκδίκασης υποθέσεων για τα εθνικά δικαστήρια και βεβαίως υπερβολικός όγκος εργασίας προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ο οποίος σίγουρα θα μπορούσε να αποφευθεί. Επομένως, σήμερα η συζήτηση αυτή είναι πολύ σημαντική και θέλω να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο. Στο βαθμό που θα εφαρμόσουμε, κυρία Επίτροπε, τα πιλωτικά προγράμματα για την κατάρτιση των δικαστών θα προβλέψουμε παράλληλα έναν ουσιαστικό μηχανισμό αξιολόγησης θα μπορέσουμε δηλαδή να δούμε αν αυτή η προσπάθεια έχει άμεσα αποτελέσματα για τους πολίτες και την καλύτερη απονομή της δικαιοσύνης. σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάσκα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το νομοθετικό περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταβάλλεται διαρκώς και αυτό ασκεί πίεση στους εισαγγελείς, τους δικαστές και τους δικηγόρους οι οποίοι χρειάζεται να εντάξουν στη δουλειά τους όλες αυτές τις αλλαγές. Γι' αυτό για εκείνους που είναι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για την εφαρμογή του δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν τη δυνατότητα διαβίου μάθησης και κατάρτισης για οικονομικούς και άλλους λόγους νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να οργανώνονται τέτοια, όταν οργανώνουν τέτοια προγράμματα να γίνεται χρήση του υπάρχοντος δικτύου εξειδικευμένων σχολών και πανεπιστημίων στα κράτη-μέλη τα οποία με κατάλληλη διαπίστευση θα παρέχουν τα αναγκαία προγράμματα κατάρτισης για το εθνικό και το ευρωπαϊκό δίκαιο στους δικαστικούς και άλλους λειτουργούς. Είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα μπορέσει μέχρι το 2020 να εκπληρώσει το στόχο της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Και τώρα θα ήθελα να παρακαλέσω την Επίτροπο εν ονόματι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απαντήσει τα ερωτήματα που ετέθησαν. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα μακρηγορήσω, η ώρα είναι προχωρημένη. Επιτρέψτε μου λοιπόν απλώς να πω ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την συμβολή σας σε αυτή τη σημαντική υπόθεση γιατί μιλάμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη δικαιοσύνης με ένα χώρο εμπιστοσύνης, για την εμπιστοσύνη απαιτείται πρωτίστως η γνώση. Είναι λοιπόν απαραίτητο να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες μαζί με τους επαγγελματίες, μαζί με τους αρμόδιους σε εθνικό επίπεδο, ώστε η γνώση να καταστεί πραγματικότητα για το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό νομικών σε όλα τα επίπεδα ευθύνη τους. Και θα ήθελα να προσθέσω και ένα άλλο στοιχείο. Την εμπιστοσύνη σημαίνει επίσης συναντήσεις, επαφές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι νομικοί μιας χώρας να μάθουν, να γνωρίσουν τους δικαστές, τους δικηγόρους, τους εισαγγελείς μιας άλλης χώρας, ώστε αν προκύψει κάποιο θέμα να γνωρίζουν σε ποιον επαγγελματία συνάδελφο θα χρειαστεί να απευθυνθούν. Αυτά τα προγράμματα που θα καθιερώσουμε λοιπόν θα είναι προγράμματα που θα φορούν το περιεχόμενο αλλά θα είναι παράλληλα και προγράμματα που θα συμβάλλουν στην αλληλογνωριμία μεταξύ των δικαστών και, και λοιπόν νομικών και λειτουργών. Ευχαριστώ. Τέλος η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12. Και τώρα ερχόμαστε εις ε, ε, ε, παρεμβάσεις διακίας ενός λεπτού. Πρώτα η κυρία Σκριντελεύσκα από το ΕΛΚ. Κύριε... Ε, ευχαριστώ κύριε